Συνεπώς, έληξε η συνεδρίαση. αυτή. Τα πρακτικά θα ε, τεθούν προς ε, έγκριση στην αρχή της ε, επόμενης συνεδρίασής μας, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Οι αποφάσεις οι σημερινές θα υποβληθούν στους αποδέκτες τους και στις αρμόδιες αρχές.